το να δώσουμε χρήματα σε κύριους κέριους τομείς όπως είναι τα προενταξιακά κεφάλαια κτλ. Αυτό θα μας βοηθήσει να δώσουμε κεφάλαια και επενδύσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το να μην δώσουμε τα 200 ε, εκατομμύρια στο Ταμείο Εγγύσεων θα σημαίνει απόσυρση της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον έξω κόσμο σε επίπεδο 5 δισεκατομμυρίων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητε να ενισχύσουμε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να ενισχύσουμε τις σχέσεις αυτής της περιοχής με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τέλος σημαντικό να υπογραμμίσω ότι αυτή η αύξηση του Ταμείου Εγγύησεων της ΕΤΕ το συνολικό ποσό στην κατηγορία 4 θα μείνει αναλύωτο. Χαίρομαι και είμαι πολύ ικανοποιημένος για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τον κύριο Κάλφιν και τους άλλους συζητητές για να φτάσουμε στο συνολικό, ε, στη συνολική οροφή 26 δισεκατομμυρίων συν ένα πρόσθετο ποσό 2 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το τωρινό επίπεδο χρηματοδότηση. Θέλω λοιπόν να ζητήσω την υποστήριξή σας για να έχουμε τα απαραίτητα ποσά μέσα στην εξωτερική εντολή της ΕΤΕ και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πείσουμε όλους τους ε, εμπλεκόμενους και κυρίως το Συμβούλιο για να μπορέσει να μην απορρίψει διαρρήδην αυτή την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά να την εξετάσει. Όπως ξέρετε η διαδικασία έγκρισης για την εντολή δανειοδότησης της ε, ΕΤΕ πρέπει να γίνει πολύ σύντομα για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικών δαπανών. Χρειαζόμαστε μια νέα τέτοια εντολή μέχρι τον Ιούνιο του 2014 το αργότερο για να μην διακοπούν οι εξωτερικές μας δράσεις. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σαφή νομική και δημοσιονομική βάση, χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Υπογραμμίζω και πάλι ότι ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με άλλους φορείς και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο σύμμαχός μας στα θέματα αυτά. Η εντολή μας δίνει μια ε, σαφή κατεύθυνση για μια συνεκτικότερη δράση και μια σωστή μόχλευση των ταμείων των κονδυλίων του προϋπολογισμού που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να υποστηρίξει επενδύσεις διατηρώντας το επιχειρηματικό της μοντέλο και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να προσθέσω ορισμένα σχόλια στην παρουσίαση που ήδη ακούσαμε. Στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και ιδιαίτερα του προπολογισμού 2014, γνωρίζουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί σε όλους τους τίτλους, σε όλα τα κεφάλαια. Ε, μία από τις δυνατότητες που θα είχαμε για να αντισταθμίσουμε αυτό το, αυτή τη μείωση, αυτές τις περικοπές, ιδιαίτερα στον τομέα της εξωτερικής δράσης, θα ήταν να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη δυνατότητα να συνεχίσει το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης τουλάχιστον να συνεχιστούν ε, τα προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για να συνεχιστεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Εάν δεν το πετύχουμε αυτό θα υπάρξουν ε, αρνητικές συνέπειες σε περιοχές τι τις οποίες εργαζόμαστε ήδη εδώ και τέσσερα χρόνια η αποτελεσματικότητα της ε, χρήσης, της μόχλευσης των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι εξαιρετικά υψηλή. Η μόχλευση 30, 30 ε, φορές σημαίνει ότι βάζουμε ένα ευρώ και καταφέρνουμε να έχουμε μια απόδοση 30 ευρώ. Δεν έχουμε τέτοιες αποδόσεις σε άλλους τομείς εύκολα. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού στο Ταμείο αυτό το εγκυοδοσίας γίνεται επί τη βάση προβλέψεων. Και γνωρίζουμε ότι κάθε αύξηση ενός δισεκατομμυρίου στη δανειοδοτική ικανότητα μεταφράζεται σε αύξηση 55 εκατομμύρια ευρώ από τον ε, προϋπολογισμό. Για το 2014 δεν θα υπάρξει ε, επίπτωση γιατί η συνεισφορά σε αυτό το έτος υπολογίζεται από τα ιστορικά στοιχεία, από τα προηγούμενα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Που σημαίνει ότι η χρηματοδοτική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Απαιδήσεων δεν θα ε, μειωθεί άμεσα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν εντωμεταξύ να βρεθούν ε, πηγές χρηματοδότησης, για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κλιγής αλλαγής θα μπορούσαν να εξευρεθούν με άλλους τρόπους. Αναζητούμε, για παράδειγμα, την ε, δυνατότητα να μεταφέρουμε πόρους από ε, το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμβάλλει. Υπάρχει επίσης μία πρόταση για αύξηση της ευελιξίας και δεδομένης της αβέβαιης ε, και εύθραυστης ε, κατάστασης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην περιοχή γενικότερα και την ε, ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και αυτό θα προσπαθήσουμε επίσης να το συζητήσουμε. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση προέκυψαν μετά από τις προτάσεις της Επιτροπής Σοφών μια σειρά προβλέψεις. Συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα πια η εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο αφορά την ε, διαφάνεια, την συμμετοχή των ενδιαφερομένων έχει βελτιωθεί και πρέπει να διατηρηθεί αυτό το κεκτημένο και τώρα πια να δούμε τα αποτελέσματα, να έχουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Και τέλος, θα έπρεπε να φροντίσουμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς την ενδιάμεση αξιολόγηση έτσι ώστε να μην ξεκινήσει αλλά να τελειώσει μέχρι το τέλος του 2014. Ε, ευελπιστούμε να τελειώσει ο τριμερής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν θα ήθελα να φτάσουμε την τελευταία ολομέλεια να συζητάμε και να χρειαστεί εκεί να εγκριθεί η εντολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στη χρηματοδότηση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί με το χρονοδιάγραμμα και να συνεργαστούμε όσο καλύτερα γίνεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να βρούμε τη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε Λαμασούρ και εγώ θέλω να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Χόιερ, τον οποίο έχω γνωρίσει στο παρελθόν όταν ήταν υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων στην Γερμανία, όταν ήμουνα και εγώ υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Κροατία και σας χαιρετίζω και πάλι στον αξίωμα σα, σας, διότι έρχομαι από μια χώρα η οποία έχει ήδη επωφεληθεί από τις εξωτερικές δανειοδοτήσεις της ΕΤΕ και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ε, ανικοδόμησης των ε, οδικών συγκοινωνιών, των σιδηροδρόμων, διάφορα σχέδια στον αγροτικό τομέα και την εκμετάλλευση του ε, φυσικού του του βιοαερίου και σίγουρα είναι σαφής προσθέμενη αξία που έχει προέλθει από τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το κύριο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι το σύνολο της δραστηριότητα της ΕΤΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνάδει απόλυτα με τις προσπάθειες της Κομισιόν, με τις προσπάθειες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία της με συνεκτικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους γεωγραφικούς χώρους που καλύπτονται από τις δραστηριότητε της ΕΤΕ και της εξωτερικής της εντολής και αυτό περιλαμβάνει την ιδιαίτερη εστίαση σε χώρες που είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες προενταξιακού χαρακτήρα και αυτό καλύπτει και την πολιτική διεύνηση και την ε, ανατολική εταιρική σχέση καθώς και την εταιρική μας σχέση με τη Μεσόγειο, όλες λοιπόν τις δραστηριότητε που βρίσκονται σε ειδικότερο πλαίσιο της δράσης ΣΕΤΕ. Εγώ εξετίμησα ιδιαίτερα τα σχόλια του φίλου μου του Ιβάιλο Κάλφιν, ο οποίος ε, έχει αναλάβει την εισηγησία για το θέμα αυτό σε σχέση με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και έχει να κάνει με το ύψος της εγκυοδοσίας για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και αυτή τη στιγμή η διαφορά βρίσκεται μεταξύ 29,5 και 25 δισεκατομμυρίων συνολικού ύψους που θα τύχει εγγύησης. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και στις μελλοντικέ δράσεις ένα ποσό αντίστοιχο αυτού του παρελθόντος και να λάβουμε υπόψη και αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος Χόιερ για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ευκαμψία. Αν λάβουμε υπόψη όμως τους περιορισμούς για τις δημοσιονομικές προοπτικές και τη Γενική Πολιτική Συμφωνία που επετεύχθη, νομίζω ότι στους επόμενους μήνες και στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να βρούμε μια συμβαστική λύση που θα παραμείνει μέσα στο γενικό πλαίσιο των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών και θα επιτρέψει οι δραστηριότητες της ΕΤΕ να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές που θέλουμε να προωθήσουμε, ιδιαίτερα χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία του κλίματος κτλ. Για όλους μας επίσης κάτι που είναι σημαντικό είναι το να ακούσουμε την ανάλυση του Προέδρου σε σχέση με τη διαδικασία χρηματοδότησης της Συρίας. Υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου τα χρήματα του προεπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα σημαντικό στόχο που είναι η παροχή εγγύησεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριο Στόλογιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. The first one is what about... Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται με την πυρηνική βιομηχανία, με τις πυρηνικές μονάδες, ό,τι έχει σχέση γενικά με την πυρηνική ενέργεια. Έχετε προγράμματα ή αιτήσει προγραμμάτων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Θεωρείτε ότι η βιομηχανία αυτή θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για τις ε, δανειοδοτήσεις της τράπεζάς σας γιατί πολλές φορές οι προτάσεις σας δεν αναφέρονται ε, στην επιλεξιμότητα της πυρηνικής βιομηχανίας. Κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με την Αρμενία στο παράρτημα 3 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιλέξιμες χώρες. Βλέπω τώρα ότι πέρασε στο παράρτημα 2 πιθανές υποψήφιες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Στολογιάν. Κυρία Μπαλτακίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι λοιπόν από τη Μάλτα, είμαι Ευρωπαία, αλλά είμαι και από τη Μεσόγειο και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω κάποιες προτάσεις από πλευρά σας και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε σχέση με το παράρτημα 1. Εξεπλάγει από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το τι περνάει στην παρούσα φάση η Μεσογειακή Περιφέρεια. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα της Αραβικής Άνοιξης, και μόνο και μόνο αυτό νομίζω πρέπει να μας κάνει να δούμε την περιοχή με διαφορετικό τρόπο. Μέσω της Αραβικής Άνοιξης έχει αλλάξει εντελώς το σενάριο για το μέλλον της περιοχής και η δική μου χώρα φυσικά έχει παίξει ένα κάποιο ρόλο. Ως εκ τούτου, εμείς στην Μάλτα παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και ήμασταν πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Λιβύη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί πιθανές ε, επιπτώσεις του τι συμβαίνει στη Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα στη Συρία. Γνωρίζουμε ότι σχεδόν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες ε, έχουν φτάσει έξω από τα σύνορα της Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει εδώ να παίξει η αλληλεγγύη, να παίξει το ρόλο ο οποίος τη αρμόζει. Και γιατί λοιπόν στην ουσία προσπαθούμε να ξεχάσουμε εμείς και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει στον Νότο. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να εγκαταλείψει τη Μεσόγειο στις σημερινές της δυσκολίες, στα διέξοδά της. Η περιφέρεια της Μεσογείου θα θα πρέπει να πάρει τα ποσά τα οποία της αναλογούσαν το 2009, δηλαδή γύρω στα 9 δις περίπου. Τα 2 τρίτα για την νότια γειτονία και το 1 τρίτο για την ανατολική γειτονία. Ε, δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε γιατί αυτό θα είναι μια παλινοδία σχετικά με τον καθορισμό των οροφών σε σχέση με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση γνωρίζουμε ότι έχουμε την σημερινή πρόταση του 20% ανά ημιπεριφέρεια, ανά Συνεπώς, οποιαδήποτε προσπάθεια ανακατανομής μέσω της ενδιάμεσης αναθεώρησης θα θεωρηθεί απειλή για το τμήμα αυτό της Μεσογείου και γι' αυτό ακριβώς το σωστό ποσοστό θα πρέπει να είναι το 10%. Πρόκειται για μια πρώτη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρήσετε αυτές τις σωστές προτάσεις σχετικά με την Νότια Μεσόγειο. Ευχαριστώ συνάδελφε. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω και εγώ δύο ερωτήσεις, οι οποίες δεν είναι το αρχικό ε, αλλά είναι σημαντικές ερωτήσεις για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή προπολογισμών. Μιλήσατε για την αύξηση κεφαλαίων που μπόρεσε να κάνει η τράπεζα αυτό τον καιρό και θα θέλαμε να έχουμε και τη δική σας αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προήλθαν από αυτή την αύξηση κεφαλαίου. Θεωρείτε ότι οι προβλέψεις που είχατε κάνει πριν από λίγους μήνες θα επαληθευτούν ή όχι και επίσης στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καταφέραμε να εδραιώσουμε την, την αρχή των project bonds σε σχέση με το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάνει μια σημαντική συμβολή. Θα μας ενδιαφέρε λοιπόν να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. και κατά πόσο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μελλοντική χρηματοδότηση. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σου καλύτερα μπορώ. Και στη συνέχεια ίσως θα μπορούσε ιδιαίτερα για τα συγκεκριμένα στοιχεία να μας βοηθήσει και η Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να βρούμε μια κάποια δημιουργικότητα όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ίσως αλλάξει και η νοοτροπία ορισμένων κρατών μελών σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Άρα, ίσως, για παράδειγμα, κάποιες πολύ σκληρές ε, απόψεις ή θέσεις που έχουν εκφραστεί σήμερα για ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ανακατανομή των κονδυλίων, θα μπορούσαν να αλλάξουν και θα μπορούσαν να γίνουν πιο φιλικές. Ε, εν τέλει πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων για αυτές τις προτάσεις και την υποστήριξη που εκφράζεται και θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζω ότι η προτεραιότητα για εκείνους που έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης δεν ταιριάζουν με την εξωτερική διάσταση. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προβάλλει μια εικόνα, να έχει μια σωστή εικόνα σε άλλους τομείς προς τα έξω, για παράδειγμα στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Και είναι επίσης σημαντικό να είναι όλο και περισσότερο ορατή, να έχει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα η δράση ε, της οικονομικής βοήθειας από την πλευρά της Ένωσης. Μπορώ να πω ότι είμαι κάπως ανακουφισμένος από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια, τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβούλιο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τις ε, προτεραιότητες και τις δράσεις της Επιτροπής. Και αυτό μας φέρνει σε μια πολύ σημαντική ερώτηση και μια σημαντική χώρα, τη Συρία. Παλαιότερα εμείς αναλαμβάναμε με δικιά μας πρωτοβουλία δράσεις προς τη Συρία και έχουμε συμβάλει σε σημαντικά επενδυτικά προγράμματα στη χώρα αυτή. Αντιληφθήκαμε όμως ότι η κατάσταση αυτή, αυτές τις επενδύσεις δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν. Πολλά χρήματα είχαν μπλοκαριστεί. Χρειάστηκε λοιπόν να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε το πρόβλημα ε, και να βρούμε μια λύση. Δεν καταφέρουμε βεβαίως να το λύσουμε στο 100%. Κάποια χρήματα που έχουν μεταφερθεί στην τράπεζα του Κατάρ μπορούμε να πούμε ότι παραμένουν στη σφαίρα επιρροής μας, αλλά εδώ χρειάζεται συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, που αναφέρατε πριν την Αρμενία για παράδειγμα, στην οποία έχουμε δραστηριότητα και θα την συνεχίσουμε, ισχύει και για άλλες χώρες της περιοχής. Πρέπει να εφαρμόσουμε παντού τα κριτήριά μας, να εξετάζουμε αν οι προϋποθέσεις που θέτουμε πληρούνται και ιδίως σε θέματα συμμόρφωσης. Αλλά πέρα από αυτό να σας διαβεβαιώσω ότι γνωρίζουμε και σεβόμαστε τις υποχρεώσεις μας στον τομέα της ανατολικής ε, γειτονίας, της πολιτικής για την ανατολική γειτονία. Και αυτό ισχύει με την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια αφοσίωση ε, και για την περιοχή της Μεσογείου. Βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα προβλήματα στη λύση των οποίων πρέπει να συμβάλλουμε εκεί. Άρα έρχονται σε πρώτη προτεραιότητα τα προγράμματα για τη, για τη Μεσόγειο. Συμμετείχα στην ε, σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας την Άνοιξη στη, στις ΗΠΑ και ήμουν ο μόνος εκπρόσωπος από ε, Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα που μπορούσε να πει ότι εμείς είχαμε αποτελέσματα. Γιατί υπάρχουν άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν να είναι πρωταθλητές στη ε, στο να υπόσχονται χρήματα, στη δέσμευση χρημάτων, αλλά εμείς καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα. Όμως το ευαίσθητο ζήτημα είναι εάν σωστή η ισορροπία ανάμεσα στη Νότο και στην Ανατολή, στη Νότια γειτονία και την Ανατολική γειτονία. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα στο οποίο εγώ δεν θα τοποθετηθώ. Πρέπει να ληφθεί η απόφαση από τους ηγέτες της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση εμείς συνεργαζόμαστε πλήρως ε, με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Φιούλε, που είναι αρμόδιος για τις πολιτικές γειτονίες. Για το ζήτημα της ε, πυρηνικής ενέργειας, αυτή τη στιγμή δεν διαβλέπω κάποιο σχετικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα που επιλέγονται, επιλέγονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη. Άρα δεν είμαι εγώ αυτός που επιλέγει. Αυτό που ήδη έχουμε κάνει όμως είναι ότι έχει γίνει μια επαναξέταση, μια αξιολόγηση της πολιτικής για την ενέργεια, στην οποία έχουμε συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και έχουμε θέσει μια σειρά κριτηρίων για το, τη χρηματοδότηση ενεργειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων παραγωγής ενέργειας. Προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία στον τομέα αυτό. Ε, για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να, πρέπει να συζητήσουμε με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο για το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη που είναι μια πολιτική απόφαση, αλλά επίσης το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και ποιος φορέας θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της σταδιακής, ε, σταδιακού κλεισίματος ε, σταθμών παραγωγή, ε, παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Δεν είναι το ζήτημα μόνο τι, ποια, τι είδους νέα εργοστάσια θα δημιουργήσουμε, τι νέους σταθμούς θα δημιουργήσουμε, αλλά τι θα κάνουμε και με τους πεπαλαιωμένους. Αυτό είναι ένας σημαντικός το ΜΕΑΣ των σταθμών παραγωγής ενέργειας και η επιλογή βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Και προς εσάς, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω ότι με βάση την αξιολόγηση που κάναμε, ορισμένες μέθοδοι που έχουμε επανελειμμένα χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, δανειοδότηση, για παράδειγμα, ε, φαίνεται να είναι αποδοτική. Ίσως είναι νωρίς για να αντιλήσουμε τα τελικά συμπεράσματα. Εν τέλει μπορεί να υπάρξουν κάποια προγράμματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι την 21η Δεκεμβρίου ή την 31η Δεκεμβρίου και ίσως το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου για παράδειγμα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια κάποια ισορροπία μεταξύ του φόρτου εργασίας που θα έχουμε στο τέλος του 2013 και στις αρχές του 2014 στο επιχειρησιακό επίπεδο. Μας διευκόλυνε σε αυτό η απόφαση που λάβατε στην εργασία με τα κρατη για την αύξηση του κεφαλαίου. Μια γενικότερη παρατήρηση. Ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργο, έργου με μεγάλη αποφασιστικότητα. Προσήλωση το θεωρούμε πολύ σημαντικό εργαλείο, αυτό το καινούριο εργαλείο και αυτά τα έργα θα πρέπει να ανταποκριθούν σε, μια, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον γιατί ανταγωνιζόμαστε με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή, έχει εξετάσει εντελεχώς αυτό το, το εγχείρημα. Και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα πριν λίγους μήνες ε, στην Ισπανία. Ή επίσης το πρόγραμμα για, σχετικό με τις offshore στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη φάση των προγραμμάτων των, ε, που θα χρηματοδοτούνται μέσω ομολόγων. Για παράδειγμα το πρόγραμμα για την αποθήκευση φυσικού αερίου θα έπρεπε κατά την άποψή μου να εγκριθεί με βάση τα παλιά κριτήρια. Θα ήταν, πιστεύω, κρίμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί σωστά από οικονομική και τεχνολογική άποψη φαίνεται πολύ καλό. θα ήταν ε, κρίμα να μην ε, στεφτεί τελικά από επιτυχία επειδή θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε σε αυτό τα νέα κριτήρια. Με χαρά λοιπόν άκουσα τις παρατηρήσεις του Πρόεδρου Μπαρόζο όταν μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πριν λίγες εβδομάδες και αναφέρθηκε στο εγχείρημα της, ε, των ε, έργου ευελπιστώ ότι αυτό θα εκφραστεί και σε ε, συγκεκριμένα βήματα με τον αρμόδιο επίτροπο. Τώρα, για ορισμένα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, ιδίω σε σχέση με τη Συρία, να δώσω τον εκπρόσωπο στην... το λόγο στον εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Μετά την απόφαση αναστολή της, αναστολής της βοήθειας προς τη Συρία, ανακοινώθηκε μια υποστήριξη της τάξης των 110 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μονάχα 81,2 που καλύπτονται από την εγγύηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μόνο η τρίτη φορά που έχει χρησιμοποιηθεί η εγγύηση και είχαμε υψηλό επίπεδο επιτυχίας όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις σε άλλες χώρες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτή την ενέργεια. Δεν ξέρουμε πόσο θα χρειαστεί σε χρονικό επίπεδο. Très bien. de... Τρέμπια λέει ο πρόεδρος, πολύ ωραία, δεν θέλει καλή στο λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κυρία μου. Εξόχως ενδιαφέροντα ήταν όλα αυτά, σας υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμά μας τώρα. Έχουμε μια σειρά από τριγωνικούς διαλόγους που προβλέπονται 16 Οκτωβρίου, 6 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου, ίσως 16, ίσως 18, ίσως 24 το βράδυ. Δεκεμβρίου δηλαδή. Αλλά για μας, μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, έχουμε καθορίσει μία προθεσμία για τις τροπολογίες 1η Οκτωβρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά διακοπή και ξεπερνάμε μέσω τώρα στις ψηφοφορίες. La Συνεχίζουμε ε, Όχι, εμείς συνεχίζουμε. Οι αντιπρόεδροι θα πάρουν τις θέσεις τους. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του Αλεξάνδρου Άλβαρο. Έχετε όλοι τον κατάλογο μπροστά σας. Όλοι εκτός από τη Γένσεν την Άννη έχετε την κάρτα. Αλεξάνδερ έχει το λόγο. Ένα πράγμα σε 30 δευτερόλεπτα και 30 δευτερόλεπτα μετά την ψηφοφορία γιατί στην παρούσα φάση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γιάν Μούλτα γιατί ανέλαβε αυτό στην προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μη θελημένης απουσίας μου τους τελευταίους μήνες. Και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βοήθησαν με πολύ επικοδομητικό τρόπο την γραμματεία και το προσωπικό και το γραφείο μου. Δεν έχω πια χρόνο και θα μου δώσετε άλλα 30 μετά την ψηφοφορία παρακαλώ. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το κατάλογο τροπολογία 28, η είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 29 της κυρία Τροτμάν. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Il Δεκτή. Οπότε καταπίπτει η 31 και η 32. Περνάμε τώρα στην 33. Η συγητής υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 34, Γιάν Μούλντερ. ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ε, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34, ηλεκτρονικός έλεγχος. Il y personnes qui ont mis la carte qui n'ont pas voté. Δύο έχουν βάλει την κάρτα αλλά δεν ψήφισαν ακόμα. Έβαλε. Ε, Η Γκούε χρησιμοποιεί πιστοτικές κάρτες για να ψηφίσει. Κοιτάξτε, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πήγα να πληρώσω το ξενοδοχείο, λέει ο πρόεδρος, με την κάρτα της κοινωνικής ασφάλισης και δεν δέχτηκαν κιόλα, περίεργο. Λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορία. 10 υπέρ, 22 κατά. Συγγνώμη, 11 υπέρ, 22 κατά ως εκ τούτου απορρίπτεται. 35. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τριάντα έξι. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 37. Λεγκρίπ. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του ιδίου του εισηγητή έχετε το κείμενο στον κατάλογό σας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 39 έχει αποσυρθεί από τον κύριο Χόμαγερ. Η 40. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, καλύπτεται η 40, η 41, η 42 καλύπτεται. 43 λοιπόν, η συγγητής υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φτάνουμε στην τροπολογία 1. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της Χολμάιερ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 της κυρίας Χολμάιερ. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Πέρα στις φοφορίες. Συνεπώς 17 υπέρ, 15 κατά. Συν 1, 16 κατά. Μηδενική αποχή, η τροπολογία 1 γίνεται δεκτή. Τώρα. Συμβιβαστική 1 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Περνάμε λοιπόν τώρα στην έξι της Μόνικα Χολμάιερ, ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο 7 της κυρίας Λεγκρή, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αν και η πλειοψηφία θα είναι η ίδια. Δύο παραμένουν εν υπνώση. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ 15 κατά δεκτή ή 8. Περνάμε στην 9. Όχι, έχει καταπέσει η 9 και η 10 έχει καταπέσει. Φτάνουμε στην 11 της κυρίας Λέγκλιπ. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται έχουμε τη 12 της Κολμάια ο εισηγητής κατά ποιοι είναι υπέρ Λοιπόν, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 12 της Χολμαϊερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος εξαφανίστηκε και δύο εξακολουθούν να κοιμούνται. Πέρα στις ψηφοφορίες 15 υπέρ και 17 κατά. 16 υπέρ 17 κατά απορρίπτεται. Αυτή ήταν η 12 της Μόνικα Χολμάγερ. Όπως έχει απορριφθεί πλέον, θα πρέπει να ψηφίσουμε την 13 της κυρίας Στροτμάνου. Η συγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 14. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Πέραση ψηφοφορίας. 18 υπέρ 13 κατά, η τροπολογία 14 γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική 2 του εισηγητή, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για μια ακόμη φορά. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Είναι αρκετά τσίμα, τσίμα. Υπάρχουν δύο ψήφοι. Αλλά τα βγάζουμε καθυστέρηση. 31 ψήφους, 18-13. 18-13 ή 18-14 εγκρίνεται. Καλύπτει τη 15, τη 16 αλλά και τη 17. Πάμε στη 18. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Οι ίδιες πλειοψηφίε. Ποιο μετράει. Θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία. Α, αλλάχ, κάποιος ξύπνησε. Πέρασε ψηφοφορίας. 19-14 η διαπλειοψηφία. 19 τροτμάν. <clears throat> Η συγκητής η συγητη υπέρ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Οχιες. Δεκτή. 20. Βιέραν φέρν και διάφοροι υπέρ. Ο εισηγητή. ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Ας ελέγξουμε και πάλι. Ας ψηφίσουμε. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν να ψηφίσουν. Καλά, συνεχίστε να προσπαθείτε. Άλλος ένας κοιμήθηκε, λέει ο πρόεδρος. Βεβαίως, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορίας. 17 υπέρ 14 κατά. Η ίδια πλειοψηφία και πάλι. Μικρή πλειοψηφία, γι' αυτό είμαι υποχρεωμένο να ελέγχω. 21 του Γκέραν. Με δύο προφορικές με προφορικές τροποποίησεις σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. την προφορική τροπολογία θα ψηφίσουμε πρώτα. Σε δύο φάσεις. Πρώτα το κείμενο με την προφορική τροπολογία. Εάν απορριφθεί το κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία. Ο εισηγητή δεν δέχεται το κείμενο με την προφορική τροποποίηση. Ψήφι υπέρ τη προφορική. Το κείμενο με την προφορική. Τα ίδια. Κατά. τα ίδια. Η ίδια πλειοψηφία. Εκτός αν θέλει κάποιος ένα έλεγχο θα κάνουμε έλεγχο αλλά αλλιώ το αφήνουμε. Το κείμενο τώρα χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Λογικό το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. 22. Η συζήτηση υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τα ίδια. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Συμβαστική 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή. Καλύπτει την 23 και την 38. 24. Ο εισηγητής την υποστηρίζει. Υπέρ κατά αποχές τα γνωστά. Λοιπόν, εγκρίνεται. 25, τα ίδια φαντάζομαι. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε την 25 και την 26 ομού. Εντάξει, υπέρ. Κατά. μικρές αλλαγές. Ελέγχουμε και για τις δύο μαζί και για την 25 αλλά και για την 26. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας προφορίας. 17 με 15. Ωραία. Δεν ήταν προφανές. Περνάμε στην 27 της Μονίκας, της Μόνικας, συγγνώμη. Η Μόνικα μάλλον ζήτησε μια χωριστή ψηφοφορία. Το κείμενο χωρίς τις λέξεις πλησίον του συνομοθέτη. Ο συγκεκριτής το υποστηρίζει. Ψήφι υπέρ. Μόνικα διστάζεις. Εδίστασες. Εδίστασες. Ο συγκεκριτής το υποστηρίζει όμως. Η Μόνικα προσπαθεί να θυμηθεί γιατί ζητάει να το υποστηρίζει. Ωραία. <clears throat> Ψήφι υπέρ πάλι. Κατά. Κανείς. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο. Χωρίς το, χωρίς το νιαγδέκο legislator. Και τώρα να προσθέσουμε τις λέξεις near the legislator. Ο είναι υπέρ. Και η Μόνικα είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Α, πρέπει να λέξω. Είναι τα ίδια πράγματα πάλι. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Near the core legislator. Μα τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό όμως. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ξυπνήσατε όλοι. Ωραία, μπράβο. 16 υπέρ, 16 κατά. 17-17, επομένως απορρίπτεται. Μαζί με αυτούς που δεν έχουμε κάρτα. Το δεύτερο τμήμα. Οπότε δεν είναι κοντά στον συνομοθέτη. Δεν ξέρω ποιο είναι ή ποιο δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κείμενο. Near the co-legislator. Τελική ψηφοφορία τώρα. έλεγχος. Ό,τι μου λένε σκιώδης κάνω εγώ. Ωραία. 28, 29, ψηφίστε, ψηφίστε. Ψηφίσαν όλοι. Οι δύο που δεν έχουν κάρτα αλληλοανερούνται. 18-15 εγκρίνεται. Η έκθεση Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Ο θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Είπα στην αρχή ότι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το λόγο για δύο δευτερόλεπτα. Τώρα που ψηφίστηκε αυτή η έκθεση, θέλω αυτούς, να ευχαριστήσω αυτούς που υπερψήφισαν, ακόμα και αν είχαν αμφιβολίες. Δεν θα σας ρωτήσω αν μπορείτε να ζητήσετε από το Γενικό Γραμματέα να δημοσιευτεί η μελέτη της Δευτέρας Σεπτεμβρίου όπου περιέχονται και μερικά από τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέραμε. Αυτό ενδιαφέρει και ευρύτερα βουλευτές εκτός της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ίσως και οι υπόλοιποι βουλευτές θα θέλουν να μπορούν να κρίνουν οι ίδιοι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αυτή η έλτιση προς το Γενικό Γραμματέα να δημοσίευσει αυτή την μελέτη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα διαβιβάσω αυτήν την ε, αίτηση. Βέβαια υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Αν υπάρχει πρόβλημα θα καλέσουμε την NSA να μας βοηθήσει. Ναι Μόνικα. να κάνω απλώς μία κρίση για το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε ψηφίσει εναντίον ορισμένων κομμάτ, κομματιών της ε, έκθεσης γιατί είχα ζητήσει από τον εισηγητή να θέσει τα νέα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση και δεν το δέχτηκε. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να το γνωρίσουν και τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου εκτός του Κοινοβουλίου. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να είχαμε τα στοιχεία αυτά τα οποία και στην κοινή γνώμη θα γίνουν γνωστά, τα ενημερωμένα στοιχεία και όχι τα παλιά στοιχεία. Και δεύτερον, είναι εν μέρη δύσκολο να προχωρούμε με μέτρα τα οποία δεν μας ε, βοηθούν ιδιαίτερα. Τα κράτη-μέλη έχουν περίπου αγνοήσει το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή των συνθηκών, ότι ψηφίζουμε πια ως Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά και δεν έδειξαν ιδιαίτερο πνεύμα συνεργασίας. Και επίσης ήταν κάπως δύσκολο να βασιστούμε στην ε, <clears throat> δίκηση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό εμείς ήμασταν εναντίον της 25ης μελέτης για τους τρεις τόπους εργασίας. Γιατί έχουμε ήδη ζητήσει 6 ή 7 εκθέσεις και λένε τα ίδια πράγματα λένε τα ίδια πράγματα, δεν χειροτερεύουν οι εκθέσει, μια χαρά είναι, αλλά λένε ακριβώ τα ίδια πράγματα ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφασίσει η δίκηση του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ για την επεξήγηση τη ε, ψήφου σα, αλλά θα πρότεινα να μην ξαναρχίσουμε την συζήτηση. Το ζήτημα είναι να έχουμε στη διάθεσή μα την Ολομέλεια, τα στοιχεία, τα αριθμητικά που χρειάζονται, έτσι ώστε να λάβουμε μια απόφαση με τα λόγω Συγχαρητήρια στον εισηγητή και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα ε, του εισηγητή Τζοβάνι Λαβία για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουν όλοι τον ε, κατάλογο με τις τροπολογίες. Κατάλογο ψηφοφορίας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη συμβιβαστική α της οποίας το κείμενο βρίσκεται στον κατάλογο υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Κανένας αποχές. Εγκρίνεται. <coughs> Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 6, κύριος Λαϊόν. Ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική β. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται και καλύπτει το, την 7. Επομένως περνάμε στην τροπολογία 8, George Lyon, υπέρ ο εισηγητής, ποιος είναι υπέρ, στο δικό μου χαρτί γράφει ότι μόνο η τροπολογία 7 καλύπτεται από την συμβιβαστική Β, λέει ο πρόεδρος. Α, ωραία. Καλύπτει και την 8 λοιπόν. Μάλιστα. Έτσι να αφηνομίζεται. Τροπολογία 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές και η γουέ Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Όλη η υπόλοιπη σελίδα τροπολογίες του κύριου Λάιον τι έχει όλες αποσύρει. Το ίδιο και η τροπολογία 3. Ο ε, εισηγητής, πάμε στην τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι, μπράβο. Πέρας ψηφοφορία, 31 υπέρ για την ακρίβεια 32. Κάνει κατά καμία αποχή συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τελειώσαμε την ψηφοφορία. Δεν υπάρχουν άλλα σημεία. Giovanni. Υπάρχει μια μεταφορά πίστοσης για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Όχι, για τα άλλα όργανα τότε. Ποιος μπορεί να πάρει τον λόγο του υπεύθυνου, η edit. Εγώ εκπροσωπώ την άποψη του Ντέρεκ. 150.000 ε, ευρώ. Γι' αυτό ζητάμε να ψηφίσετε υπέρ. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της μεταφοράς κατά αποχές. Η μεταφορά γίνεται δεκτή. Λοιπόν, μπορούμε να επανέλθουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Δίνοντας το λόγο στη Γιούτα. Για τα σημεία 11 και 12 να μας τα παρουσιάσετε από κοινού παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται και πάλι για αποκεντρωμένους φωνής ο φορέας για τους ιδιοδρόμους ΕΡΑ. Εδώ πρέπει να έχουμε μια, ζητούμε μια γνωμοδότηση σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για το πακέτο σιδηροδρόμων και τώρα η νομοθετική διαδικασία ε, γίνεται με αρμόδια ουσίας στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο φορέας σιδηροδρόμων είναι τμήμα <clears throat> αυτού του πακέτου. Πρέπει να αλλάξει ο βασικός της κανονισμός και η Κομισιόν έχει νέα καθήκοντα με τα οποία θέλει να υποφορτήσει την ΕΡΑ. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν έχει αλλάξει και γι' αυτό η πιο σημαντική μας διεκδίκηση προς την Κομισιόν και αν το πετύχουμε έχει καλό αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Η Γιούτα ομιλεί. Και για την Επιτροπή, όπως είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στο τέλος της διαδικασίας αυτής να έχουμε ένα τροποποιημένο δημοσιονομικό δελτίο. Οπότε όμως αυτό σημαίνει ότι εφόσον η ΕΡΑ, καταρχήν είναι εννοείται ότι εφόσον η ΕΡΑ έχει περισσότερα καθήκοντα, θα χρειαστεί προσωπικό περαιτέρω και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσει, να το εξετάσει η Κομισιό και να μας δώσει ένα τροποποιημένο δημοσιονομικό δελτίο. Το υπόλοιπο τμήμα των αιτήσεων έχει να κάνει με κάτι άλλο που έχουμε συζητήσει σε σχέση με, τις, ε, με τους αποκεντρωμένους φορείς, δηλαδή το οργανόγραμμα. Συμφωνούμε όλοι ότι όλοι οι αποκεντρωμένοι φορείς, ακόμα και αυτοί που έχουν νέα καθήκοντα, θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο του 1% το χρόνο ή 5% λιγότερο από το 2013 ως το 2017 να μειώσουν το προσωπικό τους. Αλλά μόνο αυτό το 1% και όχι άλλο 1% για τη λεγόμενη αναδιάταξη του προσωπικού. Αυτό το απορρίπτουμε και δεν θέλουμε να γίνει αυτό σε οποιοδήποτε αποκεντρωμένο φορέα και να υποστούν περαιτέρω μείωση 1% του προσωπικού τους. Επίσης πρέπει να τονιστεί το εξής και προς την Κομισιόν. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το 1% το οποίο έχουμε αφήσει να περάσει, να αντιμετωπίσει, να εφαρμοστεί και σε προσωπικό το οποίο συντηρείται από τα έσοδα των αποκεντρωμένων φορέων. Ξέρουμε ότι αυτοί οι φορείς οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από τέλη είναι αυτοί που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και αυτές οι επιχειρήσεις ανησυχούν τα μάλα γιατί η Κομισιόν προσπαθεί να περιορίσει το οργανόγραμμα των αρμοδίων φορέων. Γι' αυτό το έχω τονίσει στους συναδέλφους. Έχω μιλήσει με εκπροσώπους των αποκεντρωμένων αυτών φορέων και γίνεται σαφές παραδείγματος χάρη για την εναέρια κυκλοφορία. Επειδή περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια ανάκαμψη στην ε, αεροπορική, στην κατασκευή αεροσκαφών και της εναέριας κυκλοφορίας, θα υπάρξει πρόβλημα αν ο φορέας πιστοποίησης των αεροσκαφών στην κολονία δεν θα είναι σε θέση ταχαίως και αποτελεσματικά να καλύψει τις απαιτήσει της βιομηχανίας. Τότε θα αποτύχουμε. Έχουμε κάνει τόσες πολλές προσπάθειες για να αναπτύξουμε την, αυτο, την αεροπορική μας βιομηχανία και τώρα θα μας περιορίσει η Κομισιόν η οποία έχει παροπίδες και περιορισμένη όραση για τα θέματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και με την ΕΡΑ γιατί και αυτή θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο της ε, πιστοποίησης σε επίπεδο ασφαλείας. Αν λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να γίνεται με γρήγορο τρόπο και αποτελεσματικό η πιστοποίηση τότε τότε υποσκάπτουμε το έργο της. Και επομένως οι τροπολογίες μου έχουν αυτό το στόχο και επίσης <clears throat> έχουμε την άποψη, κάτι το οποίο έχει προέλθει και από την κοινή προσέγγιση στην ομάδα εργασίες, ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια, είναι πολλές φορές πολύ μικρά τα γραφεία, τα διοικητικά αυτά συμβούλια, αλλά τον έχουμε αντί για δύο, τέσσερις εκπροσώπους της Κομισιόν στα διοικητικά συμβούλια, αυτό το θεωρώ απόλυτα υπερβολικά, υπερβολικό. Όταν μιλάμε πάντα για τους αποκεντρωμένους φορείς και την αποτελεσματικότητα και τη μείωση του προσωπικού στον προϋπολογισμό τους, δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να λέμε ότι θα έχουν τέσσερις εκπροσώπους κομισιών. Έχουν να αντιμετωπίσουν το κόστος ε, διαμονής και το κόστος μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως δεν είναι <clears throat> ο κατάλληλος χώρος για να αυξήσουμε την ανάγκη χρηματοδότησή τους. Επομένως εγώ τα διαγράφω αυτά απερίφραστα. Αυτά λοιπόν για τους αποκεντρωμένους φορείς. Για την Berecom τώρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αναφέρω. Η δική μας τώρα γνωμοδότηση είναι μια έκθεση για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Πρόκειται για την αξιολόγηση της Μπέρεκ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα τα μέσα που δόθηκαν στην υπηρεσία για τις ηλεκτρονικές επι, ε, επικοινωνίες των φορέα των ρυθμιστικών αρχών αυτών. Δεν μπορούμε να δίδουμε σε ένα ρυθμιστικό φορέα κάποιες ε, αρμοδιότητες <clears throat> γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα η Μπερέκ είναι απλώς μία ε, διοίκηση που διαχειρίζεται το δίκτυο των Ευρωπαίων ρυθμιστών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είναι πάρα πολύ μικρός φορέας και έχει μονάχα 16 υπαλλήλους και περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις για ένα υποτιθέμενα ανεξάρτητο οργανισμό. Αυτά νομίζω ότι είναι βλάκιες και νομίζω ότι αποτυγχάνει αυτό το εγχείρημα αν εμείς θέλουμε να το ρυθμίσουμε έτσι, ίσως θα πρέπει να διαλύσουμε την ΜΠΕΡΕΚ και να ξαναδώσουμε πάλι τις αρμοδιότητες στην Κομισιόν να ε, διαχειρίζεται αυτό το δίκτυο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αυτό θα ήταν η πιο λογική αντιμετώπιση. Η Κομισιόν τώρα μας προτείνει μια νέα νομική βάση για να έχουμε έναν εξάρτητο φορέα ο οποίος θα λειτουργεί προς όφελος όλης της Ευρώπης και των 28 κρατών μελών και θα έχει μια άποψη για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό θα έχει νόημα αν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά όχι να έχει απλώς ένα φορέα διαχείρισης των δικτύων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που μας προτείνει η Κομισιόν δεν είναι επαρκές. και πιστεύω ότι οι αρμοδιότητες της ΜΠΕΡΑΚ πρέπει να επανέλθουν στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ο Ντομινίκ Ρικέ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια θα πω για την Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Υπηρεσία που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Να ευχαριστήσω την Ούτε για την εργασία της θα ήθελα να θυμίσω δύο στοιχεία για αυτούς που ίσως να μην τα γνωρίζουν. Το τέταρτο σιροδρομικό πακέτο, του οποίου νομίζω θα κλείσει η πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της παρούσης έντολης, ε, περιλαμβάνει δύο τμήματα, ένα τεχνικό τμήμα, στο οποίο υπάρχει, περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό στοιχείο, το οποίο είναι η δημιουργία ακριβώς η επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων εκεί θα υπάρξει συμφωνία με το, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αλλά το πακέτο αυτό το τεχνικό αλλάζει εντελώς την περίμετρο ευθύνης, την εμβέλεια ευθύνης. Πρόκειται για μία, θα έλεγα, υπηρεσία η οποία καθορίζει τα επίπεδα, ε, μελετά, ερευνά και τη ζητάμε να πιστοποιήσει όλες τις συνδρομικές επιχειρήσεις, όλο το τροχαίο υλικό, όλο το υλικό το βοηθητικό στον τομέα της ασφάλειας, να ελέγχει όλες τις εθνικές υπηρεσίες, να ελέγχει ακόμα και τα κέντρα έρευνας και διάφορες άλλες αποστολές, τις οποίες δεν θα σας κουράσω τώρα. Λοιπόν, για αυτές τις νέες αρμοδιότητες, πάνω στις οποίες συμφωνούμε βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να μειωθεί το προσωπικό μέσω μιας κάποιας αναδιάταξης του προσωπικού όπως είπε σωστά η Γιούτα και μετά να υπάρξουν 27 νέες θέσεις. Αυτό είναι ανέκδοτο. Η Επιτροπή Αναφορών, Μεταφορών συγγνώμη, που ακολουθεί την υπόθεση αυτή με προσοχή είπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η προσθήκη δημοσιονομική που είχε σχέση με τον κανονισμό αυτής της υπηρεσίας καθιστούσε ανέφικτη τη λειτουργία της υπηρεσίας σωστά. Θυμίζω ότι οι αποστολές της άπτονται της ασφάλειας του σιωδρομικού δικτύου. Λόγω ακριβώς της αποστολής που έχει η υπηρεσία αυτή και της πλήρους αναντιστοιχίας του δημοσιονομικού δελτίου με το οργανόγραμμα, οδηγούμεθα σε μια κατάσταση ιδιαίτερα θα έλεγα επικίνδυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Έχουμε να κάνουμε με ένα αδιέξοδο δημοσιονομικό ανάμεσα στο δελτίο και στις αποστολές που καλείται να αναλάβει η υπηρεσία. Αυτό που είπε η Ούτα είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν βλέπουμε τις δημοσιονομικές προβλέψεις. Λοιπόν έχουμε ένα νομικό πρόβλημα πρώτα, οικονομικό κυρίως και αν δεν υπάρξει η τροποποίηση του δελτίου του δημοσιονομικού τότε δεν θα τροποποιηθούν οι αποστολές της ΕΡΑ και θα σταματήσουμε εν τη γενέση του το τέταρτο πακέτο για, α, την, για τους ιεροδρόμους και κυρίως για την ασφάλεια τους. Πολύ καλά λέει ο Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστώ τον την εισηγήτρια και τον Ντομινίκ που μας είπαν ότι τα προβλήματα αυτά είναι σημαντικά και σε επίπεδο αρχής και σε επίπεδο πρακτικό δημοσιονομικό. Για τα δύο αυτά θέματα έχουμε κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι... όχι, δεν έχουμε. Τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν ως έχουν. Η συνεδρίασή μας είναι αυτή που είχαμε προβλέψει. Η προθεσμία 7 Οκτωβρίου, 5, ε, μάλλον 17η απογευματινή για τις τροπολογίες 17, ε, στην Ήτρη η ψηφοφορία 24 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία για την ασιοδρομική ε, υπηρεσία στις 26 στην Επιτροπή Μεταφορών Νοεμβρίου πάντα. Για το πότε θα φτάσουμε ολομέλεια δεν ξέρουμε ακόμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Περνάμε στο 10 κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Κομμουνιδά Βαλενθιάνα. Κύριε Πλένκοβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει διευμηνία στη γλώσσα μου σήμερα και γι' αυτό ε, θα παρουσιάσω την έκθεση στα αγγλικά. Πρόκειται για μία από τις εκθέσεις που κινητοποιούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αφορά τις 630 απολύσεις σε πάνω από 140 επιχειρήσεις που εντάσσονται στην περιοχή ΝΑΤΣ 2 της κοινότητας της Βαλενθιάνα. Έχουν ε, ε, δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις της περιοχής λόγω της παγκοσμιοποίησης υλικά οικοδομών, μέταλλα κτλ. Δεν είναι ανταγωνιστικές πλέον οι επιχειρήσεις αυτές, απώλεια θέσεων απασχόλησης και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στον τομέα των κοινωνικών στην ισπανική αυτή περιοχή της Βαλένθια. Τα ποσά τα οποία ε, εδώ ζητούνται είναι το, συν, το ίμιση του συνολικού κόστους της ζημίας που προκλήθηκε από τις ε, ε, συνέπειες της ε, παγκοσμιοποίησης στην περιοχή σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε άμεσα μετά από αίτημα των Ισπανικών αρχών εδώ και λίγους μήνες το μήνα Απρίλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει αυτή εδώ την πρόταση ακριβώς προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν λίγες μέρες άλλωστε στις 16 Σεπτεμβρίου και περιμένουμε τώρα την έγκριση του Κοινοβουλίου. Επί της ουσίας της κατάστασης πρόκειται για μια θα έλεγα παραδοσιακή σε εισαγωγικά απρόταση την οποία έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν από τότε που δημιουργήθηκε το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και ο εισηγητής συστήνει την έγκριση της πρότασής σας βοηθώντας ακριβώς την ένταξη ε, στην αγορά εργασίας ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων στην κοινότητα της Βαλένθια. Και ευχαριστώ και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που με βοήθησαν να συντάξω τη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών επί της εκθέσεως του συναδέλφου Πένκοβιτς καθορίζεται την 1η Οκτωβρίου, για την 1η Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία προβλέπεται στις 17 Οκτωβρίου και στην Επιτροπή μας αλλά και στην Επιτροπή Απασχόλησης που είναι συνυπεύθυνη. Καλώς επανερχόμεθα τώρα στα δημοσιονομικά. Ιάν, Ιάν Γένσεν. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε περιληπτικά την κατάσταση για το 14 μετά από την πρώτη συνάντηση των λεγόμενων διατακτών. Ε, ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχαμε πάνω από χίλιες τροπολογίες από τις διάφορες επιτροπές και από μεμονωμένους ευρωβουλευτές. Στην διάσκεψη των ε, συντονιστών ε, συζητήσαμε με τις διάφορες πολιτικές ομάδες και φαίνεται ότι καταλήγουμε σε μια συμφωνία, η γενική ε, γραμμή στο ζήτημα των πληρωμών θα είναι να μην ξεπεράσουμε το όριο, την κάναμε και τη σχετική συζήτηση σήμερα. θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με το Συμβούλιο για την κατάσταση στις πληρωμέ. Το ερώτημα παραμένει. Βεβαίω δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλα με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν πλησιάσουσαμε την Επιτροπή μας είπαν ότι μπορούμε κάτι να καταφέρουμε τώρα, αλλά απλώ μεταθέτουμε το πρόβλημα στο μέλλον. Απεστάλλει μια επιστολή τροποποιητική από την πλευρά της Επιτροπής, στην οποία καταγράφουν τη συμφωνία που επετεύχθη σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, την καινοτομία και για το, στο, το 2014 από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα σε αυτούς τους τομείς να γίνει εμπροστοβαρές. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε ένα πακέτο μεταξύ μας οι πολιτικές ομάδες στον ε, τίτλο 1α, ε, πολιτικές ανάπτυξης, η τροπιπιστική επιστολή από την ε, Επιτροπή ε, καταδεικνύει ότι σε αυτόν τον τομέα έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων, ενώ στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων έχουμε λιγότερες ε, δυνατότητες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες τρίτες ευελιξίας για να βρεθούν τα χρήματα για την Κύπρο και για το Ταμείο για του τους δεν υπάρχουν προβλήματα μετά τις ε, τροπολογία στη σχέση με την αγροτική πολιτική για την πολιτική εσωτερικών και δικαιοσύνης, καθώς επίσης και για την πολιτική για τον πολιτισμό και εκεί νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Για τον τίτλο 4 ε, υπάρχει μια συζήτηση, γιατί παραδοσιακά αυτός είναι ένας τομέας όπου το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε είναι σφιχτό, συγκεκριμένο και ως συνήθως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έλλειψη κοντιλίων για την ε, Παλαιστίνη και ε, υπάρχουν ε, προτάσεις για άλλες προτεραιότητες από τις πολιτικές ομάδες, επομένως ίσως το μέσο ευελιξίας να χρησιμοποιηθεί στον τομέα της εξωτερικής δράσης για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. Ο προϋπολογισμός που αφορά τα διοικητικά έξοδα είναι πολύ ε, περιορισμένος, φιχτός, αλλά αυτό εξαρτάται και από την έκβαση των διαφόρων υποθέσεων που εξετάζει το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο θα χάσει. Ε, ε, ιδίως όσον αφορά την υπόθεση που αφορά τις αμοιβέ 2011-2012 ε, και την ε, προσαρμογή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν να βρεθούν πόροι και αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά από τα θεσμικά όργανα και θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτό. Υπάρχει το ζήτημα του, ε, ε των ειδικών ε, εκπροσώπων αυτά τα έξοδα να μεταφερθούν από την εξωτερική πολιτική στην, ε, στα διοικητικά έξοδα, όπως θα ήταν και το λογικό. Επίσης, πολλοί βουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα πιλωτικά προγράμματα και τις σχετικές δράσεις όπου εδώ έχουμε γραμμές του προϋπολογισμού χωρίς νομική βάση. Ε, υπάρχει η δυνατότητα με αυτές να εξεταστούν, να δοκιμαστούν νέες ιδέες, αλλά επίσης ε, χρηματοδοτούνται και από εκεί ε, προγράμματα που αφορούν σε νομική βάση που ακόμα αναμένουμε να εγκριθεί. Αυτό αφορά διάφορες ομάδες, διάφορες επιτροπές. οι οροφές που έχουν τεθεί μας περιορίζουν, αλλά νομίζω ότι και εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση που να ικανοποιεί τους περισσότερους, λαμβάνοντας υπόψη μας την άποψη της Επιτροπής για το ότι είναι εφικτό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ένα έργο ίσως να καλύπτεται από άλλα προγράμματα χρηματοδοτικά. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι μάλλον προετοιμαζόμαστε, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο προετοιμασίας για την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα και το Κοινοβούλιο ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, τους κανόνες που είχαμε συμφωνήσει για την επόμενη προγραμματική περίοδο, παρόλο που δεν έχουμε εγκρίνει ακόμα το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, παρόλο που δεν το έχουμε υπερψηφίσει, εμεί ακολουθούμε του σχετικού κανόνε και θα έλεγα ότι ε, περιορίζουμε τι ε, διάφορε απαιτήσει μα σε ένα λογικό επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητές και το ε, προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό που μα βοήθησε, έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να βρεθούμε μια έναν κοινό τόπο και η τελική ψηφοφορία να μην ε, είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε, άν. Όπως είπε και η Άννα, σε σχέση με τον υπολογισμό της Κομισιόν γίνεται διαπραγμάτευση για συμβαστικές τροπολογίες για συμβασμούς μεταξύ των σχεδόν συγητών Για τα άλλα θεσμικά όργανα η Μόνικα έχει προχωρήσει πολύ, υπάρχει μια ομοφωνία για τα θέματα αυτά και μαζί με τον George Lyon έκανε μία ε, συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου η Μόνικα. Έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε προβεί σε περικοπές τριών εκατομμυρίων. Θα υπάρξουν και κάποιες ε, μεταφορές για την ε, πληροφορική και για άλλους τομείς και για πιο σύγχρονη πληροφορική θα υπάρξει μια εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων και έχουμε και κάποιες ε, άλλες περικοπές λιγότερο δημοφιλείς. Είπαμε του χρόνου ο αριθμός των... Ε, η, τα, το κόστος των αντιπροσωπιών θα κοπεί κατά 1,5 εκατομμύρια. επομένως θα έχουμε συνολικά μία μείωση κατά 7 εκατομμύρια, θα έχουμε μία συνολική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,9%. Βέβαια, δεν έχουμε το κίνδυνο να προκύψει ένα κόστος, υψηλότερο κόστος προσωπικού λόγω της πιθανής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις αποδοχές των υπαλλήλων. Ένα τμήμα λοιπόν προβλέπεται ήδη για να δούμε πώς θα καλυφθεί αυτό το πιθανό κόστος. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ελπίζουμε να γίνει πριν μέχρι το Δεκέμβριο. Η Άννη Έλτσεν έχει τονίσει ότι δεν έχει νόημα να αφαιρέσουμε όλα τα αποθεματικά για πιθανούς κινδύνους όταν ξέρουμε ότι το Δεκέμβριο είναι πιθανό να αυξηθεί το κόστος του προσωπικού δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει κάποιο περιθώριο το οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά τα, ε, όλους αυτούς τους κινδύνους με μεταφορές πιστώσεων. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο <clears throat> όπου έχει υποβληθεί και πάλι η πρόταση της Κομισιόν, το λεγόμενο abatement, οι γενικές μειώσεις του Συμβουλίου. Και υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης γιατί εκεί το κόστος ασφάλειας έχει αυξηθεί και υπάρχει και πρόβλημα με τους ειδικού εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε αυτή η συζήτηση να γίνει σε συνεργασία με την ΑΦΕΤ για να δούμε αν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα ή αν θα πρέπει να επανέλθουμε αργότερα. Και κατά τα άλλα δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα με το Συμβούλιο και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε πια κανένα περιθώριο και ενδεχομένως θα φτάσουμε στο 2014 με αδυναμία χρηματοδότησης του προϋπολογισμού, οπότε θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις να διενεργήσουμε. Δεν έχω αφιβολία, λέει ο πρόεδρος Λαμασούρ, Χαίρομαι που αυτό σας χαροποιεί. Δεν έχετε κανένα σχόλιο. <clears throat> Να κλείσουμε. Όχι, μια στιγμή. Η Άιντα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα ζητήσει το λόγο για να κάνω ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει κάτι το οποίο με ανησυχεί γιατί κανείς δεν μιλάει με καθαρό τρόπο. Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να λάβει θέση, όχι για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων, που όπως είπε η συγγήτρια είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά για τις πιστώσεις πληρωμών και εγώ ακόμα από τη Σοσιαλιστική Ομάδα πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω πάνω σε τι πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί δεν είναι σαφή τα πράγματα. Συζητήσαμε με τον Επίτροπο, κάποια πράγματα είναι σαφή, αλλά δεν είναι καθόλου. Ούτε η θέση του Συμβουλίου έχει διαμορφωθεί με σαφήνεια, γιατί λέει απλώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς που έχουμε ενώπιό μας. Δεν ξέρω τι λογαριασμούς έχουμε. Ίσως θα πρέπει να βρούμε μια άλλη στρατηγική για να εκμεύσουμε το Συμβούλιο ποια είναι η κατάσταση. Αλλά τι θα ψηφίσουμε τελικά την επόμενη εβδομάδα για τις πιστώσεις πληρωμών. Δεν ξέρω. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω αν αυτά τα οποία δεν θα πληρωθούν φέτος μπορούν να μεταφερθούν στον επόμενο χρόνο. Αλλά όταν το ρωτάμε αυτό το Συμβούλιο πει την ίσα. Δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση μάλλον γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει να έχει μια σαφή απάντηση που θα μας δώσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα ζητήσουμε περισσότερες πιστώσεις πληρωμών, θα διατηρήσουμε τα κονδύλια της Κομισιόν, του Συμβουλίου που είναι ένα δισεκατομμύριο πιο κάτω. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για τα θέματα αυτά όταν δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες για το θέμα αυτό. Πώς θα γίνει η εργασία μας. Ευχαριστώ Άιντε. Όπως μας είπες, οι προθεσμίες δεν είναι πολύ μεγάλες. Η επόμενη συνάντηση των συντονιστών προβλέπεται τη Δευτέρα από τις 4 μέχρι τις 6. Και η ψηφοφορία των τροπολογιδών θα γίνει την Τετάρτη και Πέμπτη και τις δύο ημέρες και σας παρακαλώ να είστε διαθέσιμοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μέχρι τη Δευτέρα είναι οι εισηγητές και οι σκιώδεις να συμφωνήσουν επί της στρατηγικής και να κάνουν όσο περισσότερο, όσο, να σημειώσουν όσο περισσότερη πρόοδο μπορούν και στα θέματα στρατηγικής και στα υπόλοιπα θέματα που θα συναποτελέσουν τη συμφωνία, έτσι ώστε και η γραμματεία να μπορέσει να προετοιμαστεί εγκαίρως για την ψηφοφορία. Δεν θα αποφύγουμε δεκάδες ε, ψηφοφοριών. Γι' αυτό λοιπόν όσο πιο νωρίς συμφωνήσετε τόσο το καλύτερο για όλους. Είμαι στη διάθεσή σας αν χρειαστεί για κάτι, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρετε μαζί τους. Τέλος, συμπληρωματικά με αυτά τα οποία ακούστηκαν, κάποια επιπλέον στοιχεία για τα σημεία 5, 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, ο Τζοβάνι δεν είναι μαζί μας, αλλά μπορούμε να πούμε συνοπτικά τα εξής. Το πρόβλημα των άλλων συμπληρωματικών για το 13, από τα προβλήματα αυτά, το βασικό είναι αυτό που συνδέεται με το MFF, η δεύτερη κατηγορία DAB 2 ε, που έχει γίνει DAB 8. 3,9 δις. Ο Λιθουανός Υπουργός, ο οποίος προεδρεύει, είπε ότι το Συμβούλιο θα τιμήσει τις νομικές ανηλυμένες του υποχρεώσεις. Και στο Βιλνίο, στην προηγούμενη εβδομάδα η Λιθουανική Προεδρία, υποδεχόμενη την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών, είπε πιο συγκεκριμένα και πιο θετικά αν θέλετε, ότι είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα αυτό, όπως θα ήθελε το Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν μια ανηλυμένη υποχρέωση πολύ συγκεκριμένη. Σε αυτά όμως θα προσθεθούν και άλλα θέματα, τρεις άλλες τροπολογίες, συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί, με διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το πρώτο είναι ο 6 που αφορά τα έσοδα. Για τον 6 η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παραδοσιακή λεγόμενη είδη πόροι, δηλαδή ε, τα τέλη, τα τελωνιακά, θα μειωθούν το 13 σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν γίνει πέρυσι. Αυτό υποχρεωτικά, αυτόματα αν θέλετε, μαθηματικά, θα οδηγήσει σε μια αύξηση του GNI για την αντιστάθμιση, γιατί αυτή είναι η ουσία του πόρου GNI. Καλείται να καλύψει τη μείωση των άλλων πόρων για να χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες όπως είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Αυτό στην ουσία θα οδηγήσει σε μία αύξηση κατά 2 δις 700 εκατομμύρια της συνεισφοράς GNI για το 2013. Βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι πολιτικές επιπτώσεις ε, για τους υπουργούς προϋπολογισμών. Θα χρηματοδοτήσουν 3,9 για τον ΤΑΜ 8 συν 2,7 που να ανταποκρίνονται Pas besoin de για το εγχώριο προϊόν. Λοιπόν, όλες αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν γίνει φυσικά στα πλαίσια μιας εύκολης διαπραγμάτευσης, ίσα ίσα. Στη συνέχεια έχουμε 7, Διορθωτικός 7. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ο οποίος έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των ετοιμάτων τριών χωρών για να αντισταθμιστεί το ότι οι υποσχέσεις τις οποίες τους είχε δώσει ο Βαν Ρόμπαϊ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Νύκτας της 8ης Φεβρουαρίου 2013, τη στιγμή που κατέληψε σε συμφωνία για το MFF το Συμβούλιο, δεν μπορούν να γίνουν σεβαστές. Δηλαδή μια επιταγή για τρεις χώρες. Η γραμμή στον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί επηρεάζει αρνητικά και την Βρετανική επιστροφή και έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση. Στόχος αυτού του διορθωτικού λοιπόν προϋπολογισμού είναι η ρύθμιση της συγκεκριμένου θέματος. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό συνδέεται άμεσα με το MFF, ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει εμείς να το ψηφίσουμε ταυτόχρονα με το MFF. Αν μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε λοιπόν για το MFF θα περάσει και αυτός ο συμπληρωματικός, αν δεν τότε σε αυτήν την περίπτωση θα περιμένουμε θα υπάρξει ε, τουλάχιστον και ένας ένατος διορθωτικός, ο οποίος ε, που να αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αποζημίωση των ε, ζημιών που δημιουργήθηκαν από πλημμύρες κυρίως στην Γερμανία αλλά και στην Αυστρία και ίσως και σε άλλες χώρες. 400 εκατομμύρια ευρώ. Ο μηχανισμός ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης, ο συνήθως άνω του κατοφλίου, αλλά αυτό δεν θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο γιατί πρέπει να βρούμε άλλα 400 εκατομμύρια χρηματοδότησης που θα προσθεθούν στα 3,9 δις του DAB 8 και στα 2,7 δις του DAB 6. Λοιπόν, κατά τα άλλα, και σχετικά με το δικό μας χρονοδιάγραμμα, συνάντηση των συντονιστών την επόμενη Δευτέρα, δύο ολόκληρες ημέρες για την ψηφοφορία όλων των τροπολογιών. Αν τελειώσουμε στη μια μισή μέρα τόσο το καλύτερο. Και τέλος, προς το παρόν θα παραμείνουμε λοιπόν στον στόχο να περάσουμε στην ψηφοφορία στο δεύτερο Στρασβούργο, Τετάρτη ας πούμε 23 Οκτωβρίου, πιθανώς. Και για την διοργανική συμφωνία και για τον κανονισμό MFF. Η δεσμευτικά νομική ψηφοφορία λοιπόν για το MFF. Η ψηφοφορία μας στην Ολομέλεια τον προϋπολογισμό του 14 πιθανώς και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι συνδέονται με τα προηγούμενα και σίγουρα επίσης και οι νομοθετικοί κανονισμοί που είναι σημαντικοί και που άπτονται του περιεχομένου των πολιτικών που χρηματοδοτούμε. Ενθυμίστε ότι για το MFF στο ψήφισμά μας στις αρχές Ιουλίου είχαμε διευκρινίσει ότι εμείς θα το υποβάλουμε σε ψηφοφορία με μία προϋπόθεση να εκπληρωθούν δύο όροι. Πρώτος, 3,9 του DAB8 και δεύτερος όρος να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές δυσκολίες στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης των νομοθετικών κανονισμών που έχουν δημοσιονομικές σημαντικές συνέπειες, δηλαδή ΚΑΠ και πολιτική συνοχής. Για την ε, κοινή αγροτική πολιτική μάθαμε χθε και μάλιστα και σήμερα το πρωί ότι οι τριμερείς διάλογοι έχουν ολοκληρωθεί και ότι υπάρχει μια πολιτική συμφωνία. Οπότε από αυτή την πλευρά δεν θα υπάρχει πρόβλημα από τη Γεωργία για την συνοχή. Υπάρχουν σημαντικά πολιτικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Υπάρχει το θέμα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και υπάρχει επίσης και το θέμα του, α, του αποθέματος επιδόσεων. Le sentiment que j'ai, un sentiment purement personnel, c'est que ces sujets... Αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να, σε αυτά τα δύο θέματα θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμός. Ε, έχουμε αρχίσει να συνεθίζουμε αυτού του είδους τις συναντήσεις και έχουν γίνει πολύ τριμερείς διάλογοι μέχρι τώρα και προβλέπουμε πάνω κάτω που θα καταλήξουν. Θα επαληθεύσουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες το πώς θα πάνε τα πράγματα. Ελπίζω να κλείσουν αυτά την επόμενη εβδομάδα και τότε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα δει αν θα συγκαλέσει μια ομάδα επαφής εκ νέου ή η λύση που είχε προβλέψει σε περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα, να υπάρξει μια συνάντηση κορυφής των τριών οργάνων επί τη βάση του συγκεκριμένου άρθρου της συνθήκης, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ή δεν είναι, θα δούμε. Και η διάσκεψη των Προέδρων θα επιβεβαιώσει ή θα αλλάξει την ημερομηνία που προβλέπεται για το σύνολο αυτών των ψηφοφοριών κατά τη διάρκεια της δεύτερης ολομέλειας του μηνός Οκτωβρίου. Λοιπόν αυτά Τελευταίο σημείο τώρα που παραμένει είναι το σημείο για τα buildings, για τα κτίρια. Εάν η Μόνικα θέλει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα κυρία Βελτσομποχάτα είναι επίσης ε, υπεύθυνη για το θέμα αυτό και την ευχαριστώ για τη βοήθειά της. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε στην κατάσταση ότι υπήρξε κάποια παράκαμψη των δημοσιονομικών κανονισμών από ένα ε, από ένα αποκεντρωμένο φορέα και έχει νοικιάσει ακίνητα για ποσά που ξεπέρασαν τα όρια τα οποία προβλεπόταν και έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα όπως είπε και η Γιούτα Χάουγκ για την ΕΜΠΑ, για την τραπεζική αρχή μόνο χρησιμοποιώντας το αποθεματικό μπορούμε να καλύψουμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να, κάνουμε μια, να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με κάνουν να ανατριχιάζω σε ό,τι αφορά αυτή την ε, ε, αρχή. Έχουν αρχίσει να νοικιάζουν όροφο μετά από όροφο και να τον χωρίσουν σε διάφορα τμήματα και ουσιαστικά έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Γιατί το κάνανε αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αν κάθε φορά επιτρέπουμε σε αποκεντρωμένους φορείς να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα μπατηρήσουμε τελείως. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα καλύτερο έλεγχο για τα θέματα αυτά. Στο μέλλον δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τρία τμήματα λοιπόν σε ένα κτίριο αυτού του είδους και πληρώθηκε και κάποιος ε, σύμβουλος για τα θέματα αυτά που θα, θα τους έλεγε αν θέλουν να νοικιάσουν τα άλλα δύο, τους, τους άλλο δύο ορόφους. και νομίζω ότι από την 1η Φεβρουαρίου τώρα θα ισχύει το πρώτο μίστομα, το άλλο θα αρχίσει στα μέσα Φεβρουαρίου και το τρίτο θα γίνει το Μάρτιο και το άλλο τον Αύγουστο του 2014. Ούτε μας λένε πότε θα γίνει αυτή η μίστοση. Τα ποσά που μας αναφέρθηκαν δεν αντιστοιχούν με τα ποσά στο και βλέπουμε στη σελίδα 14 να υπάρχουν και μερικά ακόμα τετραγωνικά τα οποία νοικιάστηκαν επιπλέον και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπολογιστούν αυτά τα, για τα τετραγωνικά τα πρόσθετα τα οποία αναφέρθηκαν και ζητώ από την Κομισιόν να μας δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν ο αρμόδιος υπάλληλος έχει προσπαθήσει ήδη να καταλάβει τι γίνεται, αλλά εμείς θέλουμε να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με παράκαμψη του δημοσιονομικού κανονισμού, μια εν γνώση παράκαμψη του δημοσιονομικού κανονισμού, διότι θεώρησε ο αρμόδιος της ΕΜΠΑ Τη υπηρεσίας για τα τραπεζικά θέματα ότι δεν χρειαζόταν να κάνει κάποια τέτοια ε, κοινοποίηση και νομίζω ότι και η συνεργάτη μου η οποία απασχολείται με τα θέματα αυτά έχει ήδη κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και θα θέλαμε να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει κάποια εξήγηση η τραπεζική αρχή αν δεν έχουμε λοιπόν μέχρι το Δεκέμβριο μία εξήγηση και μία ε, ανακοίνωση για αυτά τα θέματα, κινδυνεύουμε το Φεβρουάριο να νοικιαστεί το πιο ακριβό κτίριο το οποίο ποτέ έχει νοικιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεπερνάει κάθε περιθώριο που έχουμε προβλέψει για, το, για τις ε, ε, μισθώσεις, ξεπερνάει τα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό η, η μίσθωση αυτή που κάνει. Και στη Γαλλία έχουμε, είχαμε προβλήματα με τον ε, φορέα για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ από ένα αποκεντρωμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να επικρίνω αυτή την ενέργεια. Θα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ερωτήματα και πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με καμία κυβέρνηση ότι δεν μας ειδοποίησε κανείς. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ελεγχθούν όλα αυτά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την συνάδελφό μου η οποία με βοήθησε και αυτή για να διατυπώσω μια σειρά ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με τις ανεπαρκείς πληροφορίες και τις συγκεκαλυμμένες επίσης ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει για το κτίριο αυτό. Δεν είναι πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά και πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόκειται για την εταιρεία, για, την, για τον φορέα τραπεζικής εποπτείας. Ίσως λοιπόν ξέρουν κάτι περισσότερο να κάνουν σε σχέση με τα τραπεζικά θέματα και να μας βάζουν σε όλους σε δύσκολη θέση. Θα έπρεπε λοιπόν- Ακούσαμε Ακούσαμε πολλές λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι πάντα η ενημέρωσή μας ήταν καθυστερημένη και δεν μπορούσαμε να δράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Παίζαμε τη γάτα και το ποντίκι και αυτό δεν είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να μας αντιμετωπίζουν. Φοβάμαι για το τι θα γίνει στο μέλλον. Μας έχουν ήδη πει ότι έχουν ε, ε, πολλές προσφορές για μισθώσεις και θα ήθελα να ξεκινήσουν μια διαδικασία υποβολής προσφορών. Ανησυχώ λοιπόν για τις μελλοντικέ αυτές ε, καταστάσεις οι οποίες θα αρχίσουν ή μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα γιατί προβλέπεται η μετακόμιση το 2015. Δεν ξέρω λοιπόν ακριβώς τι προϋποθέσεις θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη αν θα υπάρξουν κυρώσεις, αλλά ίσως να υπάρξουν κάποιες ρήτρε πάρα πολύ περίπλοκες, έτσι ώστε στο τέλος να αναγκαστούμε να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα, επειδή εγκαταλείπουμε νωρίτερα τις εγκαταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες να σεβαστούν τους κανόνες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από την υπηρεσία αυτή να μας δώσει εγγυήσει για το σεβασμό και των πιστοτικών ρυθμίσεων. Ό,τι φαίνεται. Είμαστε απλώς εμβρόντιτοι για αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι γίνονται όλα αυτά στο Λονδίνο που είναι αστρονομικά τα νίκια είναι ακόμα χειρότερο. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε την πρόταση της Μόνικα. Θα πρέπει να δώσουμε την γνωμοδότησή μας πρώτον και δεύτερον και θα πρέπει να κάνουμε σαφή και τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται για τον προϋπολογισμό για να μπορέσει να γίνει σαφής η πίεση η οποία δημιουργείται με τον τρόπο αυτό. Λοιπόν, δεν, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που κάνουν Πώς μας αντιμετωπίζουν έτσι. Νομίζω ότι δεν κατανοούν ότι υπάρχει, αν όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του, τουλάχιστον η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για κάθε εισηγητή. Μα τι λέτε. Μου είπανε ότι υπάρχουν άτομα από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Μπορούμε να του δώσουμε το λόγο αν θέλουν να απαντήσουν. Ποιο θέλει να μιλήσει λοιπόν για τα θέματα αυτά. Παρακαλώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πέστε μας λοιπόν τι γίνεται. Το όνομά σας. Άνταμ Φάρκες, είμαι ο εκτελεστικός διευθυντής της ABA και σας ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να παρευρεθώ και με συντομία να προσπαθήσω να απαντήσω και να εξηγήσω ορισμένα από τα πραγματικά περιστατικά που βρίσκονται πίσω από αυτές τις ανησυχίες που εξέφρασε η συγγήτρια και η σκιώδη Πρώτα απ' όλα αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για να δούμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση είναι ότι όπως θα γνωρίζετε η EBA δημιουργήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2011. Η απόφαση που συνοδεύεται από την ε, απόφαση για τη χρηματοδότηση της ε, EBA ε, εγκρίθηκε καθυστερημένα και η απόφαση ήταν ότι θα κληρονομούσε όλες τις νομικές υποχρεώσεις της Επιτροπής επίπεδου 3 που ήταν, είχε την έδρα της στο Λονδίνο. Είχαμε καθυστερήσει λοιπόν την έναρξη ε, της λειτουργίας ε, της EBA. Η διοίκηση επελέγει κατά τη διάρκεια του 2011, δηλαδή όταν είχαν, είχε ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της EBA. Εγώ προσωπικά ανέλαβα καθήκοντα τον Απρίλιο του 2011. Όταν η αρχή εποπτείας για τις ε, τράπεζες ξεκίνησε να λειτουργεί, κληρονόμησε μισθωτήρια συμβόλαια για κτίρια στο Λονδίνο, στα οποία στεγαζόμαστε σήμερα. Τα εφιστάμενα λοιπόν αυτά ε, μισθωτήρια συμβόλαια, τα οποία ε, παρεδόθησαν σε εμένα προσωπικά, αφορούσαν ένα όρουφο σε έναν ουρανοξύστη και το 1 τρίτο ενός ε, κτηρίου στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Χάκου. Το 1 τρίτο λοιπόν ενός ορόφου. Αυτά τα συμβόλαια έλεγαν μέχρι το τέλος του 2014. Ναι, ναι, θα το πω και αυτό. Αυτά τα συμβόλαια είχαν υπογραφεί για μέχρι το ε, τέλος του 2014 και δεν υπάρχουν ε, ρήτρε σε περίπτωση μια ναι, ανανέωσή τους. Υπήρχε όμως μια ρήτρα break-up clause για ε, δυνατότητα να σπάσει το συμβόλαιο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι. Και αυτό που κάναμε αμέσως, σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάναμε μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για να βρούμε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα της στέγασης της ε, αρχής δεδομένου μάλιστα ότι προβλέπεται και σημαντική αύξηση του ρυθμού του προσωπικού της αρχής. Όταν ε, ανέλαβα καθήκοντα, το προσωπικό ήταν λιγότερο από 30 άτομα, σήμερα έχουμε φτάσει τα 100 ε, συμπεριλαμβάνονται ε, αποσπασμένοι, εκπαιδευόμενοι, καθώς επίσης και αρκετοί εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη που βοηθούν την αρχή. Πέρυσι, επίσης να σας πω ότι οργανώσαμε 250 συνεδριάσεις ε, με εκπροσώπους και εμπειρογνώμενες από τα κράτη-μέλη, κατά τη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες ε, άτομα έπρεπε να ε, βρεθούν σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στο γραφείο μας. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Παρεδόθησαν σε μας, κληρονομήσαμε κάποια συμβόλαια ακριβά, σε ακριβά κτίρια και έπρεπε με κάποιον τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Επιλέξαμε λοιπόν μια ε, εταιρεία συμβούλων ε, real estate και τους ζητήσαμε να βρεθεί μια λύση για να μετεγκατασταθεί τελικά η αρχή. Και να σας πω απολύτως ειλικρινά και απολύτως ανοιχτά, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση και επικοινωνήσαμε με την κυρία Χόμαγε, αλλά αυτό ε, ε, οδήγησε στο να μην έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε πλέον τη ρήτρα ε, ακύρωση του συμβολέου, το break-up clause, Επομένω χάσαμε αυτή τη δυνατότητα. Και ο λόγος που ερχόμαστε τόσο καθυστερημένα να ζητήσουμε αυτή την έγκριση είναι επειδή συνεχίζαμε τις διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με την κατάσταση. Όταν τελικά αυτή η διαπραγμάτευση για μια δεκαετή ε, μίσθωση ενός άλλου κτηρίου να βάγισε, χρειάστηκε να βρούμε μια βραχυπρόθεσμη, μια άμεση λύση. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν όλες τις ανησυχίες και τα θέματα που θέτει το Κοινοβούλιο, να τονίσω ότι από την πλευρά μας σεβόμαστε τις απόψεις του Κοινοβουλίου, το ρόλο του Κοινοβουλίου και το δημοσιονομικό κανονισμό. Τι αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε, να ε, βρούμε αφενός μια βραχυπρόθεσμη και αφετέρου μια μακροπρόθεσμη λύση. Η βραχυπρόθεσμη λύση ήταν η εξή. Να συνάψουμε μικρότερα επιμέρους συμβόλαια έτσι ώστε η έκταση των γραφείων μας, το μέγεθος των γραφείων μας, να αυξάνεται καθώς αυξάνεται το προσωπικό. Όμως όλα αυτά τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα έπρεπε να λήξουν μέχρι το τέλος του 2014, έτσι ώστε να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα στη μακροπρόθεσμη λύση στην επιλογή ενός κτηρίου για το μέλλον. Τι κάναμε λοιπόν, αρχίσαμε να μισθώνουμε άλλους ορόφους στο ίδιο κτίριο, Μερικές φορές κάποια εταιρεία έφευγε από έναν όροφο και τον νοικιάζαμε εμείς, αγοράζαμε μερικές φορές τα έπιπλα. Σε μια περίπτωση μάλιστα μιας εταιρείας που χρεοκόπησε ε, αγοράσαμε τον εξοπλισμό. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε ε, συνοστισμένοι σε αυτό το κτίριο. Το μέσο χώρος ανά άτομο ε, είναι πολύ κατώτερος του μέσου όρου στα γραφεία των ευρωπαϊκών ε, οργανισμών, ε, υπηρεσιών και όλα αυτά τα συμβόλαια λήγουν το τέλος του 2014. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν με την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, η οποία έκανε και την ενημέρωση προς την Επιτροπή Προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Επίσης ειδοποιήσαμε για την διαδικασία που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε για τη λύση του μακροπρόθεσμου προβλήματος, δηλαδή τη μίσθωση ενός κτηρίου μακροπρόθεσμα μετά το 2014. Ε, βεβαίως, λάβαμε αιτήματα για ε, διευκρίνηση γραπτός σήμερα το πρωί και σας διαβεβαιώνω ότι θα απαντήσουμε σε αυτά λεπτομερώς. Θα σας δώσουμε όλα τα στοιχεία, όλα τα αριθμητικά στοιχεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε αναλυτικά. Ελπίζω να μην καταχράστηκα το χρόνο σας ή την προσοχή σας και σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω και πάλι να επαναλάβω ότι είμαστε οποτεδήποτε μας το ζητήσετε στη διάθεσή σας, σε οποιαδήποτε συνεδρίασή σας, να έρθουμε και να εξηγήσουμε τις, τι πράξαμε και τι σκοπεύουμε να πράξουμε. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρακάμψουμε την Επιτροπή ή να κάνουμε οτιδήποτε που παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα του δημοσιονομικού κανονισμού. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Κατάλαβα ότι η βραχυπρόθεσμη λύση θα καλύψει τα προβλήματα αυτά μέχρι το τέλος του 2014. Επομένως, μέχρι το τέλος του 2014 η βραχυπρόθεσμη λύση. Εμείς Είμαστε στο τέταρτο, σχεδόν τέταρτο του 2013. Υπάρχουν κάποια εναλλακτικά κτίρια τα οποία έχετε ελέγξει όπου θέλετε να μεταφερθείτε από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Μια στιγμή κυρία Χολμάιερ. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό φαντάζομαι. δεν είσαστε ο ένας φορέας από τους δύο της κοινότητας, έχουμε άλλους 32 <clears throat> αποκεντρωμένους φορείς. Ξέρουμε ότι πρέπει να μετακομίσουν οι φορείς. Λοιπόν, πόσο έχετε προχωρήσει με αυτή τη διαδικασία για να σχεδιάσετε τη μετακίνησή σας. Το άλλο ερώτημα, <clears throat> ή μάλλον η δήλωση αυτή της κυρίας Χολμάιρ ότι όταν κάθε φορά έχετε επεκτηταθεί στο κτίριο αυτό βρήκατε πάντα αυτόν τον σύμβουλο ο οποίος έπιανε κάθε φορά και άλλες 10.000 ευρώ για τις πληροφορίες που σας έδινε και τις σύμβουλες σας. Λοιπόν, έχει νόημα αυτό, είναι λογικό. Συγγνώμη, λέει η κυρία Χολμαϊρ, πρέπει να πάρω το αεροπλάνο μου. Όταν υπάρχει η εντύπωση ότι πήραν τα έπιπλα ε, από δεύτερο χέρι, η συνολική σύμβαση μέχρι το τέλος του 2014 είναι γύρω στα 400.000 ευρώ. Το κόστος ε, μετασκευής του κτηρίου είναι 430.000. 230.000 ε, για κάποια άλλη αλλαγή και ο σύμβουλος πήρε 130.000 σε χρήματα για τις υπηρεσίες του. Και ευτυχώς που θα σταματήσουν όλα αυτά μέχρι το τέλος του 2014 και εάν φύγει κανείς πιο πριν από το τέλος του 2014 θα είναι 60.000 συν ΦΠΑ και επίσης θα υπάρχουν ποινικέ ρήτρε για, κόστος το, για το κόστος το οποίο ξεπερνά αυτά. Λοιπόν, έχετε ένα, μια ρήτα του Συμβουλίου. Σας έχει πληροφορήσει η υπηρεσία της Κομισιόν για την κατάσταση των δημοσιονομικών κανονισμών. Ήδη σας έχουν ενημερώσει για το, από το Μάιο του 2012 και σας είπαν ότι πρέπει να κάνετε κάποια κοινοποίηση και στην αρχή του προϋπολογισμού. Όλα αυτά δεν σας απαλλάσσουν από το γεγονός ότι πήρατε κάποιες αποφάσεις και κάνατε συμβάσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο για τις οποίες θα έπρεπε να μας κοινοποιήσετε και δεν έχετε απαντήσει στα ερωτήματά μας. Από το 2012 ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την κοινοποίηση. Ξέρατε ότι πρέπει να κάνετε κάτι, αλλά δεν κάνατε τίποτα. Και τώρα έχετε αφήσει να περάσει η διάρκεια της ρήτρα διακοπής του Συμβουλίου. Ξέρατε αυτό ότι από το τέλος του Ιουλίου 2012 θα μπορούσατε να είχατε κάνει αυτό το τέλος του Συμβουλίου. Λοιπόν, και τώρα μας λέτε, α το ξεχάσαμε, μα δεν μπορούμε να δουλεύουμε έτσι. Και αν αυτό το κάνει η υπηρεσία τραπεζικής εποπτείας, η οποία πρέπει να ελέγχει άλλες τράπεζες αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και εσείς οι ίδιοι είσαστε απόλυτα παράτυποι στα πράγματα αυτά, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχει σοβαρές συνέπειες. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Έχω πραγματικά πάρα πολλά ερωτήματα και έχουμε κάνει πάρα πολύ επεξεργασία για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι εδώ ήταν απαραίτητο να έχετε <clears throat> και να έχετε κοινοποιήσει όλα αυτά και τα κτίρια που έχετε νοικιάσει είναι σε τίμημα το οποίο είναι παρασάγκας πέραν των ορίων που προβλέπονται. Πρέπει κάποια στιγμή η Επιτροπή Προϋπολογισμών να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αλλά έχετε και άλλα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε τώρα. Όχι. Εντάξει. Καλά. Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της ε, Μόνικα. Θα κάνουμε μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Ναι, ναι. και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό στη διαδικασία του προπολογισμού. Ναι, Μόνικα, κάτι θέλεις να πεις ακόμα. Όχι. Αλλά δεν έχω τώρα να πω τίποτα άλλο. Μετά από αυτή την καταπληκτική παρουσίαση να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Γεια σας.